Ε, διατυπωθεί. Ερχόμαι τώρα, έχουν δημοσιευτεί, ερχόμαι τώρα στο σχέδιο εργασίας για αυτή τη βδομάδα βάσει του άρθρου 149 το τελικό σχέδιο της ε, Ολομέλειας έχει διανεμηθεί. Υπάρχει κάποια αντίρρηση. Η ομάδα του ΕΛΚ ζήτησε να υπάρξει μια συζήτηση για την ε, παράταση της έγκρισης του Glyphosate να εγγραφεί το θέμα αυτό βάσει τη έκθεση Καρίνου στην ημερήσια διάταξη. Ποιο έχει το λόγο για το θέμα αυτό? Έχετε το λόγο κύριε μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε εξ ονόματος του ΕΛΚ. Θα ήθελα να προσθέσουμε ένα σημείο για σήμερα και φυσικά εδώ αναφέρομαι στην ουσία γλυφοσάτ. Θα θέλαμε να εγγραφεί το σημείο αυτό μετά τη συζήτηση της έκθεσης του συναδέλφου Καρίμ, καθότι απασχολεί πολλούς από τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντελέ. Δεν υπάρχει μετάφραση διερμηνία στα αγγλικά. Κοιτάξτε, θέλετε να επαναλάβετε αυτό που είπατε για να το ακούσουν με μετάφραση. Ναι κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος του ΕΛΚ, όπως σας είπα, θα ήθελα να προσθεθεί η συζήτηση στην σημερινή ημερησία διάταξη, σήμερα το απόγευμα, για το θέμα, για την ουσία γλυφοσάτ. Η συζήτηση αυτή θα πρέπει να λάβει χώρα μετά τη συζήτηση της έκθεσης του συναδέλφου Καρίμ. Θα ήταν σημαντικό να συζητηθεί το θέμα αυτό στην Ολομέλεια, καθότι απασχολεί πολλούς Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Ποιο θα ήθελε να πάρει το λόγο υπέρ, υπέρ, Λάμπερτ, κύριε Πρόεδρε. Ναι, είναι κάτι που απασχολεί πολλούς Ευρωπαίους πολίτες και πιστεύω ότι μια τέτοια συζήτηση είναι πολύ σημαντική. Κατά της πρότασης ο κύριος Μπροκ. Πιστεύω κύριε Πρόεδρε ότι σίγουρα θα είναι σημαντικό το θέμα αυτό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συζητήσουμε, καθότι η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών λήγει σε μία ώρα. Δεν έχουμε λοιπόν χρόνο για να προτιμάσουμε το θέμα αυτό και να γίνει συζήτηση. Ψηφίζουμε λοιπόν. Υπέρ. Παρακαλώ πολύ, ψηφίστε υπέρ. Κατά. Μειοψηφία. Αποχές. Εγκρίνεται η πρόταση. Μα ήταν σαφές. Μπορείτε να... Μπορούμε να ελέγξουμε. Αλλά ήταν σαφέστατη η πλειοψηφία υπέρ. Αν επιμένετε όμως μπορούμε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ε, εντάξει, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Τέλος της ψηφοφορίας. 255 υπέρ, 91 κατά, 16 εποχές. Επαναλαμβάνω λοιπόν, εγκρίνεται η πρόταση. Σύμφωνα του άρθρου 100... Ε, Εντάξει, θα τεθεί το θέμα αυτό μετά την ε, έκθεση Καρύμ. Για την πέμπτη, ε, για την τρίτη, συγγνώμη, δεν έχω καμία πρόταση, για την τετάρτη πρόκειται για την απόσυρση της κυβέρνηση της Μάλτας του μέλους ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Υπάρχει κάποια άλλη πρόταση για αλλαγή στην ημερήσια διάταξη, στο σχέδιο εργασιών μας, όχι. Εγκρίνεται λοιπόν ένα δικαστικό κύριο Πιτέλα. Ναι, ήθελα επί του κανονισμού να εκφράσω μια, μια αίσθηση γιατί έχουμε σκανδαλιστεί λόγω της μεταχείρισης που επιφυλάχθηκε ε, σε αυτές τις ώρες στου, στους πρόσφυγες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ιδωμένη. Είναι απαράδεκτο και εγκληματικό να πυροβολούν ανθρώπους που προσπαθούν και αναζητούν διεθνή προστασία. Θέλω να θυμίσω ότι η ΦΥΡΟΜ είναι μια χώρα που είναι υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σας ζητώ, Πρόεδρε, να απευθύνετε μια σταθερή και αποφασιστική έκκληση στην κυβέρνηση της ΦΥΡΟΜ για να σταματήσουν αυτή την ιστορία αυτή την κατάσταση και στρέφομαι και στη Frontex για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των ε, προσφύγων. Μου λένε τώρα ότι η Αυστρία ξεκίνησε την οικοδόμηση ενός φράγμου, ενός φράχτη προληπτικού. Μα μου θυμίζει την προληπτικό πόλεμο του Μπούς. Καταστροφή. Κύριε Βέμπα. Μετά από αυτά που είπε ο κύριος Πιτέλα θα ήθελα να υπενθυμίσω όλοι θέλουμε να υπάρξει σωστή αντιμετώπιση όλων των προσφύγων αλλά θέλω να τονίσω ότι και οι ελληνικές αρχές έδωσαν δυνατότητα να στεγαστούν σε κανονικά καταλήματα οι πρόσφυγες που βρίσκονται στην ειδωμένη και αυτοί δεν θέλησαν να το αποδεχτούν. Πρέπει λοιπόν και οι πρόσφυγες να συμπεριφερθούν με τον σωστό τρόπο. Διαδικαστικό. Είχαμε ζητήσει για την Σενεγάλη ένα κατεπήγον για τον κύριο Μπίκο Μπούργκη και δεν στάθη να τον σταλεί ένα προσωπικό μήνυμα στον πρόεδρο Μπακισάλ. Ο κυρίος αυτός αναγνωρίστηκε σαν κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να αντέξει ποινή φυλάκισης και η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές πήρε την απόφαση να τον καλέσει. Κατόπιν όμως οι αρχές της Σενεγάλης τον ε, και τον φυλάκισαν. Κυρία Μπέρες, έχει συζητηθεί το θέμα αυτό πολλές φορές. Είμαι σε επαφή και με τον πρόεδρο και με την πρεσβεία της Σενεγάλης. Υπάρχει κάτι άλλο για την ημερήσια διάταξη. Όχι, μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Ξεκινάμε με το θέμα της ε, Παγκόσμιας ημέρας των Ρωμά, δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Καταρχήν θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Κυρία Επιτροπή, έχετε το λόγο. Αγαπητές κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ εξ ονόματος της Επιτροπής για την ευκαιρία που μας δίνετε σήμερα να μιλήσουμε